Ε, μάλλον, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση 200 ημερών μέχρι και ένα χρόνο. Ενώ ο νόμος λέει 90 μέρες. Αλλά τι γίνεται, εδώ έχει περάσει ένας χρόνος ήδη. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Αυτό που ζητάμε είναι να ρυθμιστούν τα πράγματα όπως πρέπει και με κυρώσεις, την επιβολή κυρώσεων. Όποιος δεν τα σέβεται αυτά να τιμωρείται και η διοίκηση και οι ιδιώτες. Εδώ, εάν ε, πας με 120 και περνάς και ένα κόκκινο φανάρι, τότε σηματοδότη θα πρέπει να τιμωρηθείς. Άρα λοιπόν να υπάρξουν κυρώσεις και σε αυτό. Εμείς συζητήσαμε με διάφορες πολιτικές ομάδες όπως και το ΕΛΚ στη Μαδρίτη και μας άκουσαν στην Βουλή την Ισπανική η Οικονομική Επιτροπή και ο κ. Φατιμ Μπάνιολ που συμφωνούν με την αναφορά μας οι πληρωμές στην Ισπανία δεν μπορούν να διατηρηθούν σε, με μια προθεσμία 200 τόσων ημερών ας πούμε δεν μπορεί να καθυστερεί τόσο πολύ η πληρωμή αυτών των υποχρέωσεων και πάμε στις τράπεζες και στις τράπεζες ούτε εκεί πετυχαίνουμε χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτόν και εδώ έχουμε και άλλο ένα νόμο. Ο νόμος ε, είναι υπέρ των μεγάλων εταιριών ε, σαν να αποτελούν ένα καρτέλ αυτές οι εταιρείε ε, και κανονίζουν σε πόσο χρονικό διάστημα θα γίνουν πληρωμές. Και με άλλη μεριά έχουμε άτομα, έχουν οικογένειες ε, οι οποίες αγνοούνται. Άρα λοιπόν αυτό προκαλεί ζημιές στις οικιακές οικονομίες, στις πιο ταπεινές με τους νόμους αυτούς. Αυτό που ζητάμε είναι αυτός ο νόμος ε, να αλλάξει. Γιατί αν περιμένουμε 4-5 χρόνια να ρυθμιστεί μια κατάσταση, όχι. Θα πρέπει να λύνεται το πρόβλημα σε ένα χρόνο το πολύ και να ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα πληρωθούν αυτά ή όχι. Και χρειάζεται να υπάρξει μια ενημέρωση και σε μηνύα βάση για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εδώ Εάν μπούμε σε μια διαδικασία δεν ξέρουμε πότε θα τελειώνουμε με αυτήν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι κάθε μήνα θα πρέπει να λέμε τι γίνεται με αυτούς που παρεμβαίνουν γιατί υπάρχουν από μικρές επιχειρήσεις ε, άτομα που συμμετέχουν θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε αυτούς τους διαγωνισμούς, σε αυτές τις προκηρύξεις να δούμε ποιοι θα πετύχουν ποιοι όλοι και λυπούμεθα και την έλλειψη χρηματοδότηση από πλευράς ε, τραπεζών και την χαμηλή ρευστότητα των οικογενειών για να αποφύγουν παρόμοιες κρίσεις. Από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχουμε ένα γενναιόδωρο, θα πρέπει να έχουμε ένα γενναιόδωρο δάνειο με επιτόκιο 1% αλλά μετά τι γίνεται όταν πάει στις τράπεζες με αυτό το χαμηλό πιτάκιο και πρέπει να απευθυνθεί στις μικρές επιχειρήσεις και στις οικογένειες, τίποτα, χάνονται αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχουν, δεν χορηγούνται. Ένα τρίτο των χρημάτων ε, των τραπεζών ε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάμε να πηγαίνει το 1 τρίτο στις, με το 1% να πηγαίνει στις μικρές επιχειρήσεις και στις οικογένειες. Μια και το παίρνουν τόσο χαμηλό να μην το κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που κάνουν οι τράπεζες είναι να καλύπτουν τις τρύπες τους, όλες αυτές τους προβληματικούς ισολογισμούς τους θα πρέπει να βοηθούν τις οικογένειες. Αυτό που κάνουν είναι δεν δημιουργούν πλούτο, δεν ε, δημιουργούν δυνατότητες. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι οικογένειες ε, υποφέρουν, δεν ξέρουν πού να πάνε για να χρηματοδοτηθούν. Και πάνε, τα χρήματα φεύγουν να αποδώσουμε για την Ισπανία αλλού. Για την Ισπανία μιλάω, πάνε στην τράπεζα τα χρήματα παραλαμβάνω. Τα χρή... Οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν. Μερικές φορές, λίγες φορές, αλλά με 8%, 10% και με πολλές πολλές εγγύησεις από πίσω. Αυτό λοιπόν ε, εδώ ε, εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Όλα αυτά δεν γίνονται να προχωράει έτσι σε οικονομία όπως τη δική μας με αυτή τη χρηματοδότηση που δεν θα πρέπει να κοστίζει τόσο. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Ε, θα πρέπει να δούμε τις εγγύσεις, ας πούμε για οικογενειακές υποθέσεις τα οι τράπεζες προχωρούν και σε κατασχέσεις και ήδη 26 κατοικίες έχουν κατασχέσει 26 ε, οικογένειες πέταξαν έξω. Για ποιο λόγο δεν ήταν φταίξιμο των οικογενειών, δεν έκαναν λάθος. Εργάστηκαν για μια εταιρεία που δεν τους πλήρωνε για την εργασία τους αυτό. Και μετά ξαφανίστηκε, πτώχευσε, έφυγε αυτή η εταιρεία. Δεν τους πλήρωσε κανείς. Δεν έχουν τα χρήματα αυτοί λοιπόν να πληρώσουν. Και έχουμε τώρα 140 ε, κατοικίες σε λίγες εβδομάδες, σε λίγους μήνες με παιδιά, με ηλικιωμένα άτομα 140 οικογένειες που θα πρέπει να φύγουν γιατί θα κατασχέσουν οι τράπεζες λόγω χρέους επειδή αυτοί δεν πληρώθηκαν χρειάζεται μια διαπραγμάτευση θα μπορούσε να δείξει μια γενεοδορία η τράπεζα και να πει εντάξει μπορείς να συνεχίσεις να ζεις στην κατοικία σου να μου πληρώσεις 200 ευρώ το μήνα και θα σε αφήσω να παραμείνεις αυτήν. Έτσι να υπάρξει μια συμφωνία για το χρέος ε, και σιγά σιγά να πληρώσεις αυτό που χρωστάς, αυτό που οφείλεις. Ε, αυτό είναι λυπηρή κατάσταση κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε. Είναι δραματική κατάσταση και όταν μιλάμε με ψηλά στελέχη του ΕΛΚ, του Λαϊκού Κόμματος, και εκείνοι υποστηρίζουν την πρόταση που υποβάλλουμε και μας υποσχέθηκαν ότι αυτός ο απέσιος νόμος θα ρυθμιστεί θα αλλάξει και θα υπάρξουν κυρώσει και όλους αυτούς που συμμετέχουν μια εναρμόνιση σχετικά με τη συμμετοχή αλλά ξέρετε σημαίνει συμμετοχή και εναρμόνιση σημαίνει ότι μπορεί να πάει ακριβώς μια ισπανική εταιρεία να πάει στο Λονδίνο και να έχει εκεί έδρα σε έναν διαγωνισμό κλπ. Και ποιος μπορεί να πάει μετά να διαμαρτυρηθεί και να πληρώνει δικηγόρο στο Λονδίνο. Υπάρχουν ήδη προηγούμενα σε αυτό. Υπάρχει μια εταιρεία που πήγε στην, ε, στο Λονδίνο για την, στην όλη διένεξη για να ρυθμιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ε, υπάρχουν και ορισμένες ομάδες πίεσης, λόμπις, σημαντικός κόσμος ε, που τα εξετάζει αυτά, τα αντιμετωπίζει αυτά. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε να ρυθμιστεί η κατάσταση και οι πολιτικοί θα πρέπει να μας βοηθήσουν, να βοηθήσουν τους ταπεινούς και όταν νομοθετούν να σκέφτονται και αυτούς, όχι τους μεγάλους και τις τράπεζες. Ο τελευταίος κανονισμός αυτού του νόμου που εγκρίθηκε στη Βουλή της 14 Σεπτεμβρίου φέτος σε όλη αυτή τη σειρά υπήρχαν και τράπεζες ε, και ε, όλο και καλύτερη θέση έχουν εκείνες και αυτό εις βάρος των ταπεινών, εις βάρος των πτωχών. Αυτό ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ που μου αφήραστε προσοχή και με ακούσατε για τόση ώρα. Σας ευχαριστούμε και τώρα η Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τον αναφέροντα για την ε, ξεκάθαρη περιγραφή της ε, κατάστασης με τις καθυστερημένες αυτές ε, πληρωμές, ποιες είναι οι επιπτώσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ποιες είναι οι επιπτώσεις στους εργαζομένους επιχειρήσεις αυτές. Όπως είπαμε και τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι ε, όντω το ζήτημα με τι καθυστερημένε πληρωμέ είναι πολύ σημαντικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στην περίοδο αυτή όπου έχουμε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε μια πρόταση από την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει το ζήτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόταση, στην Επιτροπή σας με συγχωρείτε, πρόταση η οποία έγινε νομοθεσία πλέον, εγκρίθηκε τον ε, Φεβρουάριο, πρόκειται για την ε, οδηγία 2011 κάθετος 7, όπου προβλέπονται πιο αυστηροί όροι όσον αφορά τις καθυστερημένες πληρωμές. Τα κράτη-μέλη πρέπει μέχρι το Μάρτιο 2013 να έχουν μεταφέρει την οδηγία αυτή. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη σε θελούσια βάση να κάνουν κάθε τι το δυνατό προκειμένου να υλοποιήσουν, να εφαρμόσουν τη νέα οδηγία ακόμα νωρίτερα, όσο δυνατόν νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης πρότεινε στα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι καλύτερο προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα οδηγία ακόμα και μέσα στο 2012. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ φιλόδοξη η διαδικασία αυτή και δύσκολη για τα κράτη-μέλη, ιδίω σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης και κάθε φορά που μιλάμε για καθυστερημένες πληρωμές δεν θα πρέπει να, μιλάμε, να ξεχνάμε το μέγεθος του φαινομένου αυτού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία πέρυσι. Οι ζημίες εξαιτία των μη πληρωμών ή καθυστερημένων πληρωμών ήταν 320 ε, ε, δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μεταφερθεί γρήγορα αυτή η νέα οδηγία στα κράτη-μέλη συστήσαμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη. Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας αυτής έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο και έγινε και μια εκστρατεία πληροφόρησης, ενημέρωσης, προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά η οδηγία αυτή σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και στο δικαστικό σύστημα, δηλαδή και οι δικαστές πρέπει να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτοί θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ε, ομοιογενώς την οδηγία αυτή παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένα την κατάσταση στην Ισπανία. Το είπαμε και στο παρελθόν και το ξαναλέμε και τώρα ότι η υπαριθμό νομοθεσία 3 του 2004 στην Ισπανία μετέφερε τις διατάξεις της υφιστάμενης οδηγίας όσον αφορά τις καθυστερημένες πληρωμές. Έκτοτε είδαμε ότι στις 5 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, μία νέα νομοθεσία εγκρίθηκε στην Ισπανία, η οποία εφαρμόζει διατάξεις της νέας οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές και πρέπει να πούμε ότι η νέα μεταρρύθμιση της ισπανικής νομοθεσίας προβλέπει μία εναρμόνιση όχι μόνο για τις δημόσιες αρχές οι οποίες συναλλάσσονται με τον ιδιωτικό τομέα αλλά αναφέρεται επίσης αυτή μεταρρύθμιση και στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών φορέων. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα λοιπόν που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς θέλουμε να έχουμε από τα κράτη-μέλη τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταφέρουμε και εμείς να δούμε ότι όντως εφαρμόζεται σωστά η οδηγία αυτή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριο Σιτουργκάης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Άκουσα την Επιτροπή. Ε, νομίζουμε ότι δίνει δίκιο στον αναφερόμενο και στα όσα αναφέρονται στην παρουσίαση, στα στοιχεία αυτά του αναφέροντα, ο οποίος και έλαβε το λόγο. Με εκπλήσει γιατί στην τοποθέτηση της Επιτροπής ε, αφήνει στην άκρη τα πράγματα, δεν μπαίνει σε βάθος, σε λεπτομέρειες. Ε, θα ήθελα να ξέρω κάτι περισσότερο. Μήπως θα μπορούσε να μας ενημερώσει για αυτή την ε, παρακολούθηση, όχι μόνο στην Ισπανία και σε υπόλοιπες 27 χώρες, ε, σε όλες τις 27 χώρες, για μια οδηγία και να πούμε τι γίνεται εδώ στην Επιτροπή για το θέμα αυτό. Τι ακριβώς ε, κάνουμε εκτός από την ακρόαση του Φεβρουαρίου που είπατε ότι θα οργανωθεί. Τι ακριβώς πέρα από αυτά στις διάφορες χώρες για παρόμοιο θέμα. Θα θέλαμε αυτό το σχόλιο γιατί θα ήταν σημαντικό να το έχουμε στην Επιτροπή μας. Εάν οργανωθεί αυτή η ακρόαση το Φεβρουάριο θα είναι ανοιχτή κλειστή ακρόαση, κλειστή ακρόαση. Τι θα γίνει, πώς θα τα πούν αυτά πράγματα. Κανονικά οι αναφερόντες θα είναι και οι για να τα ε, ακούσουν αυτά. Θα είναι κλειστό όμως, θα είναι ανοιχτό, να μπορούν να παραστούν. Τι θα γίνει, όπως και για άλλου που έχουν ε, παρόμοια πράγματα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε πώς θα γίνουν αυτά. Όλα αυτά τα αφήνουμε ανοιχτά. και θα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα, να πρέπει να μπορούμε να τα συζητήσουμε μπροστά στους ενδιαφερόμενους και στην Επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα σε αυτές τις ακροάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μουνίτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα, ο οποίος μας περιέγραψε την υπόθεση αυτή Αναφερόμαστε εδώ σε μια ισπανική υπόθεση, αλλά μπορούσε αστικά να υφίσταται σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Συνεπώς θα πρέπει να εμπλακούμε άμεσα, χρειαζόμαστε τη νέα αυτή νομοθεσία στο παρελθόν είχα και εγώ συμμετάσχει στην άμεση επεξεργασία της οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Επομένως, η όλη διαδικασία αναθεώρησης αυτή τη φορά θεωρώ ότι είναι πολύ αργή. Στην Ισπανία υπάρχει εθνική νομοθεσία, η οποία θεωρητικά εφαρμόζει την υφιστάμενη οδηγία του 2004 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών και στη συνέχεια εγκρίθηκε μια νέα ισπανική νομοθεσία η οποία εφαρμόζει τη νέα κοινοτική νομοθεσία για το ζήτημα. Καταλαβαίνω όμω απόλυτα το πόσο υποφέρουν οι οικογένειες των ανθρώπων αυτών εξαιτία των καθυστερήσεων αυτών των πληρωμών. Και νομίζω ότι ε, ένα μερίδιο της ευθύνης φέρουν και οι ισπανικές ε, τράπεζες, οι οποίες λαμβάνουν μεγάλα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια δανείζουν τα ποσά αυτά με υψηλούς ε, τόκους, με υψηλά επιτόκια, με συγχωρείτε. Υποτίθεται ότι ζούμε σε μια χώρα κοινωνικής πρόνοιας και κανονικά θα έπρεπε να επιτρέπουμε στις ε, οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη από περισσότερα χρήματα να έχουν πρόσβαση στον δανεισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι η κοινοτική νομοθεσία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρω και θα πρέπει και η Ισπανική κυβέρνηση να, να ενσωματώσει αυτή τη νέα νομοθεσία από το 2013 όπως προβλέπεται, αλλά όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και την κατάσταση των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. με συνάφο Χιμένεθ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον αναφέροντα. Είμαστε στο πλευρά του και σε όλους εκείνους που έκαναν παρόμοιες αναφορές ε, με αυτές τις απαιτήσει και στην Ισπανία με λαϊκή βάση και επίσης μπορούμε να πούμε ότι και στον προηγούμενο για όλη αυτή την ε, απελπισία τους ε, και θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό, χειροκροτώ αυτή την ιδέα που θα πρέπει να προωθήσουμε. Όπως είπαμε είναι δύσκολα τα πράγματα αυτά, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να ε, μην, να μην περάσει πολύ χρονικό διάστημα γιατί εδώ βλέπουμε ακούει τη φωνή των πολιτών και ανησυχούν και είναι καλό που ακούσαμε την ε, χρονιά το 2012, αλλά θα ήθελα να χαιρετήσω και την Επιτροφή Εμπειρογνωμόνων, όπως είπε και ο Σιτουργκάης, και πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση θα προσπαθήσει τέλος πάντων ε, να κάνει οτιδήποτε πέρασε από το χέρι της για την οδηγία αυτή γρήγορα, αποτελεσματικά και θα πρέπει να δούμε και το πρόβλημα της τράπεζας εντάξει εγώ δεν μπορώ να σας διαβεώσω και να σας χαροποιήσω αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε δηλαδή. Κρίμα, είναι απίστευτο που δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά στις επιχειρήσεις και τις μικρές και στις οικογένειες, αυτά τα χρήματα που δεν φτάνουν στους πολίτες και θεωρώ όπως και οι υπόλοιποι λόγο ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή μέχρι να έχουμε αυτή την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει το θέμα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ ο αναφέρον έχει το λόγο για να μας πει αυτά τα τελευταία. Αυτό με, την, με τις προθεσμίες, όλα αυτά είναι κολπάκια τώρα εδώ, τι γίνεται. Υπάρχει αυτό το παράδοξο, για να τηρήσει κανείς τον νόμο θα πρέπει να υπάρξει ένα έγγραφο που να λέει ότι πληρωμείται σε 90 μέρες το παίρνει η τράπεζα και λέει όχι δεν θα πληρώσω τώρα, θα σου δώσω ένα άλλο έγγραφο για άλλες 90 μέρες. Άρα λοιπόν συνολικά αυτοί έχουν 90 90 180 μέρες. Άρα υπάρχουν και άλλα χειρότερα. Εντάξει υπάρχουν κολπάκια έτσι νόμιμα που παρακάμπτουν τον νόμο αλλά και τον ζημιώνουν. Γι' αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε αυτό ιδιαίτερα προσεκτική και ένα μητρό να υπάρχει για αποδείξει πληρωμών τιμολόγια ότι αυτοί πλήρωσαν τόσες μέρες μετά. Εντάξει, σ' αρέσει αυτή η εργασία. Εντάξει, με πληρώνεις αν με πληρώσεις με 180 μέρες μετά, τι γίνεται εδώ από την ε, η ε, ημερομηνία αυτή και πέρα ισχύουν αυτές οι 90 μέρες. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Αυτό που είπε και πριν. Ένα κανονισμός που να επιβάλλει κυρώσεις. Αν κάτι άλλο γίνεται, τότε τιμωρείται. Όποιος δεν πληρώνει, να τιμωρείται. Όποιος το κάνει έτσι ελαφρά την καρδία. Θα πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους. Και την επόμενη φορά, όταν έχουμε μια υπογραφή για πληρωμή μέσα σε μια προθεσμία, να είναι πραγματικό. Έτσι, να ισχύσει. Ευχαριστώ. Γεια. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπόδειξη ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και το τελευταίο σημείο που έδειξε ο αναφέροντας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα ήθελα να είμαστε πολύ πρακτικοί εδώ. Έχουμε δύο διαφορετικά ως τύπους ανθρώπων ή εταιριών, αν θέλετε, που πρέπει να πληρωθούν. Αν κάποιο, για παράδειγμα, έχει παραγγείλει κάτι και κάτι πάει στραβά, αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό έχει αντίκτυπο στις πληρωμές. Αλλά μετά υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ότι δεν θα πληρώσουν παρόλο που έχουν παραγγείλει. Αυτό είναι εγκληματικό. Για αυτούς που αποφασίζουν εκ των προτέρων ότι δεν θα πληρώσουν, ε, δεν θα πάρετε ούτε τόκους ούτε τίποτα από αυτούς. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει τόκος υπερημερίας, γιατί δεν θα το πληρώσουν ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μια εγκληματική πράξη, το να μην εξοφλήσει ένα λογαριασμό. Από την άλλη πλευρά, όταν κάποιο περιμένει να πληρωθεί για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι εγκληματικό. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε ένα μητρό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη Γερμανία πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η καλύτερη λύση θα ήταν, για παράδειγμα, να είχαμε ένα είδος μητρώου. Η ιδανική λύση ε, είναι βέβαια μόλις παραγγείλεις ε, ένα σακάκι να το πληρώσεις ε, στο χρόνο που πρέπει να το πληρώσεις. Υπάρχουν νομικά προβλήματα και πολλές φορές οι νομικοί εμπειρογνώμονες δυσκολεύονται να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Είναι πολύ ε, περήφανοι για τους κανονισμούς που υπάρχουν, αλλά αυτοί που αποφασίσαν ότι δεν θα πληρώσουν, θα πληρώσουν ποτέ. Θα πρέπει να κάνουμε μια ακρόαση, να δούμε, να εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα, διότι πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι είναι αθώοι, τελικά μπλέκονται σε τεράστιες δυσκολίες και τελικά αναγκάζονται να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιάρπ. Η αναφορά αυτή αποτέλεσε ένα πολύ καλό εργαλείο για να προκολουθήσουμε σε κάθε βήμα την εξέλιξη στην Επιτροπή για τόσο λεπτό θέμα. Αν δείτε αυτό το φάκελο για την, επι... για την αναφορά, από το 2010 μέχρι τώρα έχουμε κάθε ενημέρωση της Επιτροπής για την αλλαγή της οδηγίας που εγκρίθηκε και μάλιστα οριστικά τον Ιανουάριο του 2011. Νομίζω ότι εντάσσεται στην διαλογική. Θα πρέπει να δεχτούμε την πρόταση των συναδέλφων που πήραν το λόγο και να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και να μπορέσουμε στους πολίτες μας να προσφέρουμε πρόσβαση σε αυτούς που, σε αυτούς που Υποβάλλονται τις αναφορές τους για μας, να μπορέσουν να συμμετάσχουν και στην ακρόαση, να παραστούν στην ακρόαση για όλα αυτά και για την οδηγία. Είναι δραματική η κατάσταση και ελπίζουμε και εμεί με την εργασία μας να δώσουμε μια όθηση ώστε αυτή η οδηγία που νομίζω ότι συγκλίνει προς αυτά που λέει ο αναφέρονα και άλλοι πολίτες αυτά να τεθούν όσο γίνεται καλύτερα και μάλιστα όσο γίνεται πιο σύντομα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον αναφέροντα, ευχαριστώ και τους συναδέλφους και περνάμε τώρα στην επόμενη το είχαμε πει σήμερα το πρωί, στα 15 και 16 οι αναφορές αυτές αναβάλλονται για άλλη συνάντηση. Περνάμε λοιπόν στην 17 η 1655 του 2010 σχετικά με την προσβασιμότητα και τον καθολικό σχεδιασμό για τα άτομα με αναπηρία είναι απόν ο αναφέρον και έχει το λόγο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής, η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η αναφορά αναφορά την, ε, ε, την, τον την έλλειψη προσβασιμότητας στον σχεδιασμό για τα άτομα με αναπηρία. Ε, υπάρχει μια οδηγία για την εισαγωγή ελαχίστων απαιτήσεων και έτσι όταν χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τότε η προσβασιμότητα και τα κριτήρια θα πρέπει να τηρούνται. Η Κομισιόν θέλει να υποδείξει ότι υπάρχει η ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που έχει ε, υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 19 ε, από τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντική αυτή για την προσβασιμότητα, διότι ορίζει την, την προσβασιμότητα και την κάνει νομικά δεσμευτικά. δεσμευτική. Η προσβασιμότητα σημαίνει ότι άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση επίση όρη σε φυσικό περιβάλλον, στην ε, μεταφορά, στην πληροφόρηση και την επικοινωνία. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι η Λετωνία έχει κυρώσει αυτή την σύμβαση, για αυτό θα πρέπει να τηρεί τις ε, διατάξεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ε, κυρώσει ε, αυτή την σύμβαση και δεσμεύεται σε αυτήν. Όταν πρόκειται περί προσβασιμότητας, οι αρμοδιότητες συγκρίζονται στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν την κύρια αρμοδιότητα να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα. Ωστόσο υπάρχουν τομείς προσβασιμότητας που εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την προσβασιμότητα. Η Κομισιόν στο παρελθόν και συνεχίζει τώρα να υποστηρίζει την προσβασιμότητα. Γι' αυτό ε, αποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία που ξεκίνησε το 2010 για μια Ευρώπη ελεύθερη για όλους, χωρίς φραγμούς και η προσβασιμότητα είναι ο στόχος αυτής της στρατηγικής και μια, ένας από τους, μια από τις κύριες ε, αξίες. Η προσβασιμότητα είναι μια ένα προαπαιτούμενο για τα άτομα με αναπηρίες για να ασκούν τα δικαιώματά τους ε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και σύμφωνα με τον χαρτί των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην στρατηγική για τις αναπηρίες αναφέρεται ότι η Κομισιόν θα ετοιμάσει ένα ε, μια πράξη, ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα. Αυτή τη στιγμή είναι σε προετοιμασία αυτή η πράξη. Ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα αγαθών και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει έτσι και πρέπει να στηρίζεται ε, σε μια ε, προσέγγιση καθολικού σχεδιασμού για να υπάρχει εναρμόνιση των προτύπων προσβασιμότητας. Ε, η Κομισιόν εδώ και καιρό έχει ε, εντολές τυποποίησης, για παράδειγμα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, στο δομημένο περιβάλλον και αυτά τα πρότυπα θα διευκολύνουν την υλοποίηση του νομού περί προσβασιμότητας. Δεν θέλω να επισέλθω στις λεπτομέρειες ε, του νόμου περί προσβασιμότητας, αλλά θα ήθελα να σας πω μερικά από τα στάδια στην προπαρασκευαστική διαδικασία. Πριν από δύο εβδομάδες ε, υπογράψαμε, κλείσαμε την σύμβαση για την προπαρασκευαστική μελέτη. Θα συλλεχθούν στοιχεία για το κόστος και τα ωφέλη αυτής της ε, μελέτης. Ε, η Κομισιόν επίσης ε, θα κάνει ένα ευρωβαρόμετρο για να κατανοήσουμε πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες το θέμα της προσβασιμότητας και την περασμένη Δευτέρα η Κομισιόν ξεκίνησε μια ευρεία διαβούλευση με όλους τους συμμετόχους, άτομα με αναπηρίες αλλά και επιχειρήσεις και παροχούς υπηρεσιών για να έχουμε τα σχόλιά τους σχετικά με το νόμο περί προσβασιμότητας. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για την προσβασιμότητα. Ο αναφέρον ζητά να έχει, υπάρχει οδηγία. Το 2013 ελπίζουμε ότι αυτό το δεσμευτικό μέτρο θα βρεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου για να μπορείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι επίσης για την ε, η προσβασιμότητα ηλεκτρονική, διότι έχουμε αυτό το ευρύ νόμο περί προσβασιμότητας που είναι υπό προετοιμασία, αλλά έχουμε και πρωτοβουλίες σε άλλα θέματα. Το ψηφιακό θεματολόγιο ε, λέει ότι θα υπάρχει ε, ανάπτυξη ε, και πρόταση για να διασφαλίσουμε ότι οι στοθέσεις δημοσίου τομέα είναι προσβάσιμες. Αυτά προετοιμάζεται τώρα η μελέτη ε, επιπτώσεων. Τώρα, σχετικά με την χρηματοδότηση στην προσβασιμότητα, ο προγραμματισμός ε, με την χρήση των διαθρωτικών ταμείων γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Αλλά στο κανονισμό για τα διαθρωτικά ταμεία, όπως έχει αυτή τη στιγμή, αλλά και στην αναθεώρηση και η Κομισιόν πρότεινε την αναθεώρηση να γίνει αυτό το χρόνο, ε, λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται ε, και χτίζονται θα ε, λάβουν υπόψη τους τα κριτήρια προσβασιμότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι δυνατόν να μιλήσω λετωνικά. Δεν υπάρχει καμπίνα διερμηνίας ε, στη γλώσσα μου, άρα μάλλον δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου. Από όσο γνωρίζω όμως μεταδίδεται μέσω του ίντερνετ ζωντανά αυτή η συνεδρία. ενδεχομένως και πολίτες από τη χώρα μου θα ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση θα μιλήσω στα αγγλικά. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τόσο την Πρόεδρο όσο και την ε, Γραμματεία που συμπεριέλαβαν το σημείο αυτό στη μερίσια διάταξη. Και μάλιστα συμπεριλήφθη η αναφορά αυτή πολύ γρήγορα από την ημερομηνία κατά την οποία υπευλήθη. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σαφή απάντηση που έδωσε σε αυτή την αναφορά. Και ελπίζω ότι η αναφορά αυτή θα παραμείνει ανοιχτή. Από ό,τι ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όντως υπάρχουν πολλές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών. Εμείς όμως βρισκόμαστε εδώ σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, και χρειαζόμαστε περισσότερες δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Και το αίτημα αυτό για πιο αυστηρά πρότυπα και πιο αυστηρές οδηγίες έχει υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, αναμένουμε τώρα την αντίδραση του Συμβουλίου όσον αφορά αυτό το νέο σχέδιο για την οριζόντια οδηγία για τη μη διάκριση για διάφορους λόγους συμπεριλαμβανομένης και της αναπηρίας. Σε εφαρμογή τις εργασίες που γίνεται προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αναφορά αυτή. Από όσο γνωρίζω από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, τα πράγματα κινούνται γύρω από αυτό το ζήτημα των μη διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως μας είπε ότι υπάρχει και μία σημαντική χρηματοδοτική συμβολή από τα κράτη-μέλη. Προτείνω λοιπόν να διατηρήσει η Επιτροπή μας ανοιχτή αυτή την αφορά Ελπίζω να έχουμε σύντομα μία σαφή απάντηση από το Συμβούλιο και να μας δοθούν και περισσότερες πληροφορίες για το πώς κινούνται τα πράγματα εκεί, δηλαδή πώς εξελίσσονται οι συζητήσεις για τη νέα οδηγία. Αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή λετονική αναφορά. Εφόσον όμως το ζήτημα αυτό εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο και εφόσον αναμένεται και μία αντίδραση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να υποβάλω μία πρόταση για τη δική μας την Επιτροπή, προς εσάς κυρία Πρόεδρε, ενδεχομένως να υποβάλουμε εμείς μία έκθεση πρωτοβουλίας βασιζόμενοι απλώς σε αυτή την αναφορά και θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης. Και αυτό να γίνει βάσει απλώς των αναφορών αυτών που αφορούν τις μη διακρίσεις για λόγους αναπηρίας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό όταν θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και από τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Αυτή είναι η πρόταση τουλάχιστον που κάνω σήμερα όσον αφορά το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις από τη Λετωνία που κατέβαλαν πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να υποβληθεί μια κοινή αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ρήγα, η οποία έδωσε έναυσμα θέλετε στην αναφορά αυτή καθότι ε, ουσιαστικά από εκεί πέρα ξεκίνησε η ομαδική αυτή συλλογική αναφορά η οποία έφτασε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προς Ευρωπαϊκό Γιάρ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον αναφέροντα. Έχουμε εδώ πέρα ένα πρόβλημα το οποίο διονύζεται, το αντιμετωπίζουμε συστηματικά και νομίζω ότι όντως θα πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά ιδίως γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή συμβαίνουν πολλά πράγματα στα πλαίσια της Επιτροπής μας και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Έχουμε το, το νέο σχέδιο διατάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι και η αναφορά αυτή θα μπορούσε να εμπλουτίσει την όλη εργασία που γίνεται αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ λοιπόν με την προλαλή σας. Νομίζω ότι αυτή την απόφαση πρέπει να, σε αυτή την απόφαση πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ τους συναδελφούς και τους αναφέροντες. Από την Επιτροπή ακούσαμε ότι είναι ανοιχτή η κατάσταση, χρειάζεται να το προσέξουμε όλα αυτά. Θα μας προσφέρουν και στοιχεία τη συζήτηση, κάτι που είναι σημαντικό και να συμμετάσχουμε, επαναλαμβάνω, να αφαιθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά για να μπορέσουμε να επιδράσουμε. Και αυτό που είχαμε πει και υπενθυμίζω σήμερα, η Επιτροπή μας έχει αναλάβει παρόμοια εργασία στη σύνταξη εγγράφου για τη νέα στρατηγική για τις ειδικέ ανάγκες και τις αναπηρίες και στη σημερινή φάση των εργασιών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την ε, πρόταση της συναδελφού Ζανόκα στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών να τα προωθήσουμε αυτά για να αποφασίσουν εάν ή όχι χρειάζεται μια παρόμοια έκθεση πρωτοβουλίας. όπως το τόνισε και η συνάδελφος Τζανόκα, δυστυχώς δεν έχουμε πολυπληθή παρουσία. Απόψε θα το δούμε στους συντονιστές, πάντως αυτό καταγράφεται στα πρακτικά, τα όσα μας είπε δηλαδή, για να πάμε παρακάτω. 10 746 του 2008 από ένα πολίτη εστονική ηθαγένεια σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγει σε εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των προσώπων με προσδιορίστη LT ε, Redding ηθαγένεια που ζουν στην Εσθενία. Ο αναφέρον είναι απόν, το λόγο έχει η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Η αναφορά αυτή του 2008 σχετίζεται με την κατάσταση που υφίσταται στην Εστονία, όπου τα άτομα με απροσδιόριστη ηθαγένεια δεν έχουν το δικαίωμα εκλέγην σε εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύμφωνα με τον αναφέροντα αυτό οδηγεί σε ένα δημοκρατικό έλλειμμα σε αυτή τη χώρα. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει μία ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με, το, με την αναφορά αυτή. Η αναφορά αυτή άνοιξε εκ νέου από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, η ανάλυση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη κατάσταση δεν έχει τροποποιηθεί. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή αποψή μας από την προηγούμενη μας ανακοίνωση, στην οποία είχαμε πει ότι όσον αφορά την ε, συμμετοχή ατόμων που δεν είναι υπήκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές, το ζήτημα αυτό δεν καλύπτεται από την κοινοτική νομοθεσία. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια γνωρίζει ότι η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα λεπτή και ευαίσθητη και γνωρίζει ότι έχουν εκφραστεί σχετικές ανησυχίες σε διάφορα φόρα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινοτική νομοθεσία καλύπτει μόνο την συμμετοχή των υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκλογές. Όπως γνωρίζετε, η κοινοτική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους υπήκους Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές και στις δημοτικές εκλογές ανεξάρτητα από το κράτο μέλος στο οποίο κατοικούν. Να προσθέσω κάτι ακόμα όμως. Έχουμε την περίπτωση Έμανες Βίνκα, εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Αρούμπα. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, το 10, επανέλαβε ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να ρυθμίσουν τις εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες δεν εναρμονίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν ποια είναι τα άτομα αυτά τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές αυτές, σε ευρωπαϊκές εκλογές. Όσο έχει λοιπόν σήμερα η κατάσταση, εναπόκειται στα κράτη-μέλη να καθορίσουν ποια είναι τα άτομα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Συνεπώς, Μόνο σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τζανόκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας παρουσίασε την τοποθέτησή της. που δυστυχώς δεν έχει τροποποιηθεί, μολονότι έχουν υποβληθεί πολλές αναφορές για το ζήτημα αυτό. Στο παρελθόν, όταν συζητήσαμε άλλες σχετικές αναφορές, είχαμε πει ότι υπάρχει ε, μια σημαντική αντίφαση θέσεων, τοποθετήσεων όσον αφορά το υπο, ε, υποεξέταση ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε την κατάσταση αυτή όπου ουσιαστικά δεν δίνανται χιλιάδες πολίτες στην Λετωνία, στην Εστονία να συμμετέχουν σε εκλογές και λέγεται πολλές φορές ότι η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί παραβίαση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της επιστολής της Vivian Redding λέει ότι έχει λάβει γνώση της κατάστασης και ότι δεν αποτελεί όμως παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Εγώ θεωρώ ότι αποτελεί παραβίαση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να σε επενθυμίσω ότι τα άτομα αυτά με απροσδιόριστη ηθαγένεια που ζουν στην ε, Εστονία, στη Λετωνία, καθώς επίσης και στη Σλοβενία είναι άτομα τα οποία είναι άτομα με απροσδιόριστη ηθαγένεια ακριβώς επειδή εξαφανίστηκε το κράτος από το οποίο προέρχονται. Η Σοβιετική Ένωση για τη Λετωνία και την Εστονία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γεκοσλαβίας για τους πολίτες που εντοπίζονται τώρα στη Σλοβενία. Επομένως τα άτομα αυτά γίνανε απάτριδες, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις προέρχονταν από συγκεκριμένε χώρες ή είχαν γεννηθεί στις χώρες που κατοικούν ή τουλάχιστον ζούσαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στις χώρες αυτές. Και αυτό διαφοροποιεί την κατάστασή τους από τους ξένους. Οι αλλοδαποί, οι οποίοι ζουν μονίμως σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούνται μετανάστες από τρίτες χώρες και έχουν ως εκ τούτου το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές στις δικές τους χώρες, δηλαδή εκεί πέρα που είναι υπήκοοι. Ενώ τα άτομα αυτά στα οποία αναφέρομαι δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε καμία απολύτως εκλογή, σε καμία περίπτωση εθνικών εκλογών, αλλά ούτε σε τοπικές εκλογές μπορούν να συμμετέχουν, ούτε σε ευρωπαϊκές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επομένω, δεν έχει δίκιο όταν λέει ότι ε, αυτοί που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εκλογές υπάγονται σε εθνική νομοθεσία. Υπάγονται και στην κοινοτική νομοθεσία, εφόσον υπάρχουν οι κοινοτικοί κανονισμοί που λένε ότι οποιοδήποτε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιοδήποτε πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές εκλογές σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Συνεπώς, οι κοινοτικοί αυτοί κανονισμοί υπερβαίνουν τους εθνικούς κανονισμούς. Τα κράτη-μέλη αποδέχονται αυτή την κοινοτική νομοθεσία και ουσιαστικά βλέπουμε μέσω της ισχύω αυτής κοινοτικής νομοθεσίας πόσο άδικη είναι η κατάσταση τελικά, γιατί υπάρχουν πολίτες από ένα κράτος μέλος μπορούν να πάνε σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ένωσης και να συμμετέχουν στις εκλογές. Ενώ ένας μόνιμος κάτοικος αυτής της χώρας δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. ότι το άτομο αυτό μπορεί να διαμένει για πάρα πολλά χρόνια, είναι κάτοικος δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Πολύ συχνά έχουμε παιδιά ανθρώπων οι οποίοι φτάσανε σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό έχει συμβεί στη Λετωνία και την Εστονία. Τώρα, στην επιστολή της Βιβιάν Ρέντινγκ λέγεται... Μάλλον παρέχονται κάποιες γενικές αναφορές στο ζήτημα της ενσωμάτωσης, της ένταξης. Η ενσωμάτωση όμως είναι ένας άλλος απλός όρος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Και είναι συζητήσιμο τελικά το τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ενσωμάτωση. Για τη συγκεκριμένη αναφορά, ενσωμάτωση σημαίνει απόκτηση της υπηκότητας, πολιτογράφηση. Αν όμως έχουμε ένα άτομο το οποίο είχε στο παρελθόν την υπηκότητα ενός, άλλους, ενός άλλου κράτους που έχει εξαφανιστεί πλέον, θα πρέπει και το άτομο αυτό να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε εκλογές, γιατί στη διαφορετική περίπτωση έχουμε μία πλήρη παραβίαση των συμβάσεων της, των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και ο χάρτη των δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπουν για αυτό το δικαίωμα του εκλέγην. Η δικιά μου μητέρα, η οποία πέθανε φέτο, θεωρείται και αυτή άτομο με απροσδιόριστη ηθαγένεια. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, όλες αυτές οι αναφορές που γίνονται γενικόλογα στην ενσωμάτωση δεν μπορούν να αλλάξουν στην πράξη τα πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς από τους οποίους αφαιρούμε τα βασικά τους δικαιώματα. Ουσιαστικά δεν φταίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Το μόνο το οποίο έγινε ότι εξαφανίστηκε το κράτος από το οποίο προέρχονται και πολλέ φορέ στη θέση του κράτου αυτού προέλευσή του που έχει εξαφανιστεί έχει προκύψει ένα νέο κράτο το οποίο του ζητά πολλέ φορέ να περάσουν από διάφορε εξετάσει προτού του δοθεί η, η υπηκότητα του νέου αυτού κράτου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω παρόλα αυτά την κυρία Ρέντινγκ, η οποία στην επιστολή της λέει και την παραθέτω ότι ε, αν τεθεί κάποιο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως η μη διακρίσεις, ε, τότε στην περίπτωση αυτή θα αναλάβω δράση. Στην περίπτωση αυτή έχουμε διάκριση, έχουμε διακριτική μεταχείριση. Επομένως χρειαζόμαστε για αυτό το λόγο παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταπολεμηθεί αυτή η διακριτική μεταχείριση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει η Επιτροπή Αναφορών να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Ξέρετε ότι θα ψηφίσουμε, τουλάχιστον ελπίζω ότι θα ψηφίσουμε τον Φεβρουάριο, αν δεν υπάρχει περαιτέρω παράταση. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή, μάλλον θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά μέχρι να εγκριθεί τουλάχιστον η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή η υποεξέταση αυτή τη στιγμή έκθεση όσον αφορά την ηθαγένεια και τα σχετικά ζητήματα. Ο κύριο Γιάρ. Ναι, και εγώ πρέπει να πω δεν είμαι ειδικό στον τομέα. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα βρίσκεται σε κάποιο άλλο επίπεδο μάλλον άλλο από αυτό που μας έχει παρουσιάσει ε, ο αναφέρον. Δηλαδή τα, άτομα που δεν έχουν ε, ηθαγένεια ευρωπαϊκή δεν έχουν δικαιώματα το εκλέγην. Πρέπει να πούμε εδώ ότι έχουμε υπηκόους που έγιναν απάτριδες διότι χάθηκε το ίδιο τους το κράτος και ξαφνικά δεν έχουν ε, δικαιώματα ψήφου. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι καθόλου ειδικό στο θέμα αυτό, αλλά ε, πρέπει, ε, υποθέτω, να έχουν την υπηκότητα κάποιου από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αν κάποιο έχει καταστεί απατρίς γιατί δεν υπήρχε το κράτος του ή εξαφανίστηκε, ε, δεν πρέπει να είναι τόσο εύκολο να αιτηθεί την υπηκότητα κάποιου άλλου κράτους μέλους. Το θέμα της αρχής του ότι μόνο υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετέχουν στις ε, ε, εκλογές. Ε, δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτή τη θέση, αλλά θα πρέπει να ίσως να συζητήσουμε αυτές τις ειδικέ περιπτώσεις. Άρα το πρόβλημα δεν είναι περισσότερο στη δεύτερη πτυχή που ανέλησα, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, αλλά ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν ευρωπαϊκή υπηκότητα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Ίσως αυτό είναι, να είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Έμειναν πολύ λίγα άτομα στην αίθουσα. Αν αυτή τη δεύτερη πτυχή της ανάλυσης μου είναι ορθή, θα πρέπει να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή, διότι εκεί μπορεί να υπάρχει θέμα διάκρισης. Αν είναι συζητάμε για την αρχή ε, τη συμμετοχή σε εκλογές. Αυτό δεν είναι θέμα διακρίσεων και είναι σαφές. Αυτή θα είναι και η γενική άποψη της ομάδας μου. Εάν είσαι άπατρης, αν έχει εξαφανιστεί το κράτος, πώς μπορείς να αποκτήσεις μια νέα υπηκότητα. Αυτό είναι το ζήτημα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, είχαμε την επανένωση. Και αμέσως ε, οι άνθρωποι βρήκαν, ε, πήραν νέε υπηκότητε. Αλλά νομίζω το, το ερώτημα μου στην Κομισιόν είναι σε αυτές τις χώρες είναι αδύνατον, είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία, ε, μήπως εκεί υπάρχουν διακρίσεις ε, σε επιπτώσει όπου κάποιο άτομο γεννήθηκε σε ένα κράτος, αλλά το κράτος στη συνέχεια διαλύθηκε. Ε, είναι αδύνατον για αυτά τα άτομα να αιτηθούν μιας νέας υπηκότητας. Γιατί δεν γίνεται. το τελευταίο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι δυνατόν ή δεν είναι δυνατόν. Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι ακόμα και αν η Τατιανά Σανούκα συνεχίζει να συνεχίζει τα γεγονότα ότι στην Εστονία και στη Λετωνία είναι παρόμοια τα πράγματα. Δεν είναι. Ξέρουμε ότι στη Λετωνία, ναι, υπάρχουν ε, άτομα χωρίς ε, ηθαγένεια που δεν μπορούν να ψηφίσουν στην Εστονία. Αυτό ε, ισχύει εδώ και 15 χρόνια μπορούν να ψηφίζουν. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα δύο κράτη-μέλη ξανά, ποτέ. Και τέλος, τα γεγονότα. Στην περίπτωση της Λετωνίας και της Εστονίας, η Σοβιετική Ένωση εξαφανίστηκε. Όπως είπε η Τατιάνα, η εξαφάνιση του κράτους ε, ε, οδήγησε σε άτομα χωρίς πατρίδα. Έπρεπε είτε να επιλέξουν τη ρωσική ηθαγένεια ή την λετονική ή την εσθονική. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Στην περίπτωση της Εσθονίας είχαμε, είμαστε ε, μειοψηφία στη χώρα μας μετά από κατοχή από τις ε, σταλινικές ε, δυνάμεις που ήταν παράνομη η κατοχή αυτή. Τώρα το 1 τρίτο μη εσθονών ατόμων βρίσκονται εκεί, αλλά το 2003, πριν από 8 χρόνια δηλαδή περίπου, άτομα με απροσδιόριστη ηθαγένεια που δεν είχαν αποφασίσει είτε να πάρουν τη ρωσική είτε την εστωνική ήταν το 12% του πληθυσμού. Σήμερα είναι στο 6,9%. Άρα οι διαδικασίες συνεχίζονται ε, ο κόσμος αποφασίζει, παίρνει τις αποφάσεις του και εμείς το σεβόμαστε αυτό. Και αυτό αποδεικνύει πόσο καλά είναι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πήραμε χρηματοδοτική βοήθεια για να κάνουμε όλα αυτά τα προγράμματα προσαρμογής. Δεν νομίζω ότι ε, πρέπει να συζητήσουμε του κατά πόσο υπάρχουν άτομα που δεν έχουν ευρωπαϊκή υπηκότητα και κατά πόσο θα πρέπει να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Είναι σαφές. Ε, οι Βραζιλιάνοι που ζουν στην Πορτογαλία ή οι ε, Πακιστανοί που ζουν στο Λονδίνο δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ε, Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, αν υπάρχει οποιαδήποτε διάκριση εναντί τόμων που ε, έχουν γίνει απάτητες λόγω εξαφάνισης κράτους, θα πρέπει να το διαρευνήσουμε. Και εγώ με τα χαράς ε, μπορώ να σας δώσω οποιαδήποτε στοιχεία για να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει διάκριση στην Εσθονία και παρόλο που δεν γνωρίζω καλά τους ε, γείτονές μου, νομίζω και στη Λετωνία τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Και τέλος, να σας πω και κάτι, το οποίο μπορεί να είναι νέος. Η Σοβιετική Ένωση, αυτή καθ' αυτή, ήταν παράνομο κράτος, διότι δεν δημιουργήθηκε με τη βούληση των ανθρώπων, αλλά με την τρομοκρατία των Πολσεβίκων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ζανόκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ να απαντήσω την ερώτηση που ετέθηκε. Ναι, ευχαριστώ και ταντια για τα ξεκάθαρά σας λόγια. οι Πακιστανοί λοιπόν που ήρθαν στο Λονδίνο ή πήγαν στο Λονδίνο ή οπουδήποτε αλλού στη Μεγάλη Βρετανία σε άλλα κράτη-μέλη, αυτοί είναι μετανάστες και έχουν την υπηκότητα του Πακιστάν διατηρούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές του κράτους της πικότητάς τους. Δεν στερούνται καθόλου του δικαιώματος ψήφου και ασκούν αυτό το δικαίωμα στο κράτος της υπηκότητάς τους. Όταν μεταβούν σε ένα άλλο κράτος μέλος γνωρίζουν ότι θα είναι κάτοικοι ενός άλλου κράτους μέλους. Στην περίπτωση τώρα ενός κράτους το οποίο εξαφανίζεται στην επικράτεια στην οποία ασκούσε την κυριαρχία του, αν αναφερόμαστε στο τι έγινε στην αρχή του 20ου αιώνα, τότε υπήρχε κάποιο άλλο κράτος, η Ρωσική Αυτοκρατορία που είχε την επικράτεια των εδαφών. Μπορούμε να πάμε και στο 19ο αιώνα, αν θέλουμε να εξετάσουμε όλη την Ευρώπη. Το γεωπολιτικό χάρτη της Ευρώπης του 19ου αιώνα. Μπορούμε να πάμε και στους Αμπισβούργους και λοιπά. Το πρόβλημα είναι εδώ μιλάμε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα συγκεκριμένο άτομο, τη Μαξίμ, Ρέβα, που συνέταξε αυτή την αναφορά και δεν έχει δικαίωμα εκλέγην για 20 χρόνια τώρα. Ναι, μιλάμε συγκεκριμένα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτού του συγκεκριμένου ατόμου. Γεννήθηκε στην Εσθονία και στερείται αυτού του δικαιώματος να συμμετέχει σε εκλογές, οποιασδήποτε εκλογές ούτε σε τοπικές. Έχει ένα μάλλον ε, ε, ενεργό ε, δικαίωμα να ψηφίζει στις δημοτικές εκλογές μόνο, αλλά όχι να εκλέγεται. Αυτή είναι παραβίαση ενός δικαιώματος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Και η διαδικασία συνεχίζεται, τα πράγματα άλλαξαν τα ποσοστά άλλαξαν. Ναι, αυτά είναι γενικά λόγια. Εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός συγκεκριμένου ατόμου το οποίο παραβιάζονται τα δικαιώματα. Αυτό συνένταξε την αναφορά και ε, την οποία υπέγραψαν κάποιες χιλιάδες ατόμων. Δεν ε, μπορείτε να υποκαθιστάτε αυτούς τους ανθρώπους συντάχθηκε αυτή η αναφορά από κάποιον το οποίο παραβιάζονται τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα. Δεν μπορείτε εσείς ε, να ε, αναφέρεστε... Εσείς ε, είστε μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, έχετε, έχετε δικαιώματα. Ο κύριος Ρέβα όμως στερείται αυτών των δικαιωμάτων εδώ και τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους Ο Σναφος Γιάρ, ναι. Ε, ναι. Δεν είναι όμως αυτό το περισσότερο σημαντικό. Οι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να ε, ψηφίζουν σε ευρωπαϊκές σε δεν είναι μια διάκριση, είναι ένα κεκτημένο. Τώρα θα πρέπει να δούμε το εξής. Οι αναφέροντες θα ήθελα να, αποκτήσουν την, θέλουν να αποκτήσουν την εστονική ηθαγένεια και τους την αρνούνται. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε. Αν τους την αρνηθούν είναι διάκριση. Αν τους πούνε «Ναι, εντάξει γεννήθηκες εδώ αλλά δεν σου παραγώ την ηθαγένεια, δεν σου την ηθαγένεια, τότε αυτό αποτελεί διάκριση. Και πάνω σε αυτό χρειάζεται να δούμε τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν περιπτώσεις που σε μερικού για ορισμένους λόγους που δεν καταλαβαίνουμε και ιδιαίτερα, τους αρνήθηκαν την ηθαγένεια. Επαναλαμβάνω πάντω, δεν είμαι ειδικό στο θέμα, αλλά το ότι μόνο οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν να ψηφίσουν, αυτό, πρόκειται, αυτό είναι ακεκτημένο, έτσι, και όχι διάκριση. Τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε. Τώρα και μια αφελής κάπως ερώτηση ο αναφέρον δεν επιθυμεί την ηθογένεια, την ιστονική είτε δεν του την χορηγούν. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ελέγξω για να είμαι 110% σίγουρος για το συγκεκριμένο αυτό άτομο που ονομάζεται Μάξιμ Ρέβα, ο οποίος έχει την ηλικία μου. Το άτομο λοιπόν αυτό από το 1993 έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση για οποιαδήποτε υπηκότητα, εστονική, ρωσική ή οποιαδήποτε άλλη. Και τώρα, πόσο γνωρίζω, έκανε αίτηση προκειμένου να γίνει κάτοικος, υπήκος μάλλον, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του παραχωρήθηκε το δικαίωμα αυτό. Επομένως είναι Ρώσος υπήκος και αυτή είναι η επιλογή του. Για ποιο το λόγο λοιπόν παραπονιέται ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές εκλογές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Όκεν. κυρία Όκεν. Δεν μπορώ εγώ να σας δώσω την απάντηση και δεν ξέρω τις ακριβείς λεπτομέρειες. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής, μια ερώτηση μάλλον. Η Εστονία έχει εφαρμόσει τη σύμβαση των απάτριδων γιατί ξέρετε ότι έγινε ολόκληρη μάχη στη Δανία. Υπήρχαν πολλοί απάτριδες Παλαιστίνοι που είχαν γεννηθεί στην Δανία και σύμφωνα με τη σύμβαση θα έπρεπε να λάβουν την υπηκότητα εφόσον το επιθυμούσαν. Αρκεί βέβαια να μην είχε εξεκραβωθεί υψηλό επίπεδο κλιματικότητας, αυτό λεγότανε. Έγινε ολόκληρη διαμάχη από την προηγούμενη κυβέρνηση στην Δανία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μας πει η συνάδελφος αν στην Εστονία τουλάχιστον υπάρχει κάτι τέτοιο. Και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ρώσου υπηκόου. Δεν ξέρω αν η σύμβαση αυτή συγκεκριμένη έχει εφαρμοστεί τελικά στην Εστονία. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει επικυρωθεί, αλλά πρέπει να το ελέγξω. Να αναφέρω με σύμβαση αυτή. Μα κοιτάξτε, εγώ ξέρω σίγουρα ότι η Εστονία δεν την έχει εφαρμόσει. Στην περίπτωση εκείνη που έχει καταργηθεί, αν θέλετε, η χώρα προέλευση. Η σύμβαση αυτή κανονικά προβλέπει ότι τα άτομα τα οποία προέρχονται από τη χώρα αυτή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν απάτριδες. Πρέπει να πάρουν την υπηκότητα της χώρας στην οποία μένουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Ε, σας ευχαριστώ. Συναδελφοί, αλλά να σας πω ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερα ευρύ περιθώριο δράσης, όπως φαίνεται άλλωστε από τα κείμενα, τα έγγραφα που εξετάσαμε. Για την έκθεση αυτή έχουμε προσπαθήσει από το 2008 ήδη και υπάρχει από τον υπογράφοντα μια αναφορά ακριβώς ότι δεν μπορεί να δει πού ακριβώς είμαστε αρμόδιοι και αν είμαστε αρμόδιοι σε αυτό εδώ για την Ιθαγένεια. Με την αφορά όμως ευαισθητοποιήθηκαν οι, συν, οι συνάδελφοι, εντάξει όχι επισήμως, ε, ίσως με την πρόταση κλεισίματος αυτός της αναφοράς. Μήπως θα μπορούσαμε να παροτρύνουμε την αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας, ε, να την παροτρύνουμε για να δει τι θα κάνει με την ανιγνώριση την εθνική όσον αφορά την ηθαγένεια. Αλλά δεν νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι έχουμε και κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα στην οποία θα μπορούσαμε να βασίσουμε τη συνέχιση της ε, συζήτησης. Προτείνω λοιπόν να κλείσει εδώ η αναφορά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Τελειώσαμε έτσι με τα διάφορα σημεία στην ημερήσια διάταξη, στο πρώτο μέρος της ημερήσιας διάταξης για το τμήμα Β αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν. Είναι αντίθετη συνάδελφος Μάγερ για τη 773, 670, 834 του 2005 και το πλάνο συναδέλφου Μάγερ του 2009 και την 445 του 2011 από πλάσια Τουργκάη. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να έχει ζητήσει εξαίρεση για τις υπόλοιπες. Για τις υπόλοιπες εντάξει ισχύει αυτό που προτείνει η Επιτροπή. Ολοκληρώνονται έτσι οι εργασίες μας και πάλι να ευχηθώ στους συναδέλφους και να πω καλό χρόνο σε όλους. Καλή χρονιά θα σας δούμε σε λίγες εβδομάδες την επόμενη χρονιά.